Ας συνεχίσουμε παρακαλώ. Περνάμε στην τελευταία φάση με τα συμπεράσματα των εργαστηρίων μας, των τριών ομάδων εργασίας που συστήσαμε. Και μετά θα ακούσουμε και τους ομιλητές. Όποιος θέλει το λόγο μπορεί να τον λάβει. Όπως σας είπα, συνεδρίασαν ταυτόχρονα τρία workshop, τρεις ομάδες εργασίας ε, με διαφορετικά θέματα, η κάθε μία. Όλοι παραπονιούνται ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο, ότι ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα για τα τρία εργαστήρια. Και φυσικά όλοι θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στις επιμέρους συζητήσεις και να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Αλλά γυράσκω ήδη δασκόμενο. Κάθε χρόνο μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Και του χρόνου που επίσης θα έχουμε κάποια αντίστοιχη εκδήλωση επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν όσοι το επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Θα ακούσουμε τώρα τα συμπεράσματα των τριών ομάδων εργασία, των τριών εργαστηρίων που είχαμε. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ερνέστ Ουρτασούν, που είναι ο εισηγητής στο πρώτο εργαστήριο για τη βία κατά των ε, προσφύγων γυναικών. Κύριε Ουρτασούν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους, όλες και όλους ε, που ήρθατε. Είμαι ο εισηγητής ε, του πρώτου εργαστηρίου, της πρώτης ομάδας εργασίας. Αν ξεχάσω κάτι, μπορούν τα μέλη που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας να με συμπληρώσουν. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με συμμετοχή ευρωβουλευτών, εθνικών βουλευτών και μελών της κοινωνίας των πολιτών. Είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τις ε, οργανώσεις των γυναικών, να εφαρμόσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να καταργηθεί η ατιμορρασία κατά των αυτούργων ε, της βίας βάρος των γυναικών. Είχαμε πρόταση μιας συναδέλφου από την Κύπρο. Επίσης, ε, οι συμμετέχοντες μας φώτισαν για τις νομικές πτυχές των νομοθεσιών των χωρών μελών. Η Ρουμανία μας έφερε μια χαρμό συνείδηση ότι η Ρουμανία επιτέλους θα εφαρμόσει την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολης και μια συνάδελφος από την Ελλάδα μας ε, παρουσίασε την εμπειρία της Ελλάδα με 800.000 ε, με 8.000 μάλλον ε, πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών ε, και των παιδιών, γιατί πολλές φορές είναι εγκαταλειμμένοι στη μοίρα τους ε, και η μόνη έδειξη και χειρονομία ελληνική δίνεται από τοπικό πληθυσμό. Μεγάλο πρόβλημα. Συνάδελφος από την Πορτογαλία επίσης μας είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα σωστά νομικά μέσα που έχουμε από τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη και τις ε, σωστές νομοθετικές διατάξεις, αλλά αυτά υπάρχουν στα χαρτιά και στην πράξη δεν εφαρμόζονται σε πολλές χώρες μέλη, κάτι που επηρεάζει φυσικά αρνητικά την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών. Και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Μία συνάδελφος από τη Γαλλία μας είπε για την κατάσταση στη Γαλλία, όπου στον Οργανισμό για τους Πρόσφυγες έχουμε ειδική ομάδα που ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες η Julie Ward, ευρωβουλευτής, έθιξε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη συζήτησή μας. Είπε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες σήμερα δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Ακόμη και ευρωβουλευτές ε, τα αγνοούν. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Τζάκλιν Πρίνς μας παρουσίασε την άποψη της Προεδρίας, της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Και τέλος, α, ακούσαμε μια κοινωνική λειτουργό, την Μίνα Τζαφ, πολύ σημαντική παρέμβαση. Μας εξήγησε η κυρία Τζαφ ότι είχε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Αφγανές που έφταναν με τα παιδιά τους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί έπρεπε να μείνουν στο υπεθρό ή σε ανοιχτό κατάλημα που μοιράζονταν τον ίδιο χώρο με άνδρες, αντιμετώπισαν εκδηλώσεις βίας και σεξουαλικής βίας. Μερικές φορές οργανώθηκαν οι γυναίκες και κρατούσαν βάρδια για να προστατευτούν από τους άνδρες που βρίσκονταν στο ίδιο κατάλημα. Είχαμε τέτοια παραδείγματα που τα ακούσαμε. Επίσης η κυρία Ρέιλι από την Επιτροπή για τις Γυναίκες Πρόσφυγες μας είπε το 55% των προσφύγων που πραγματοποιούν το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη είναι γυναίκες ή κορίτσια και ε, υπόκειται στον κίνδυνο βιασμού, σεξουαλικής βίας, αναγκαστικής, ε, αναγκαστικού γάμου, ηλωτίας, ε, μερικές φορές οι σπαντρεύουν στις χώρες τους. Πολλές φορές χρησιμοποιούν το σεξ ως συναλλακτικό μέσο για να πληρώσουν για το ταξίδι ή για τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Και πολύ σωστά μας είπε η κυρία Ρέιλι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επαρκής προστασία αυτών των γυναικών ούτε στα κέντρα υποδοχής, ούτε στα κέντρα διέλευσης. Αυτό το συζητήσαμε και στην έκθεση. Η κυρία Ρέιλι επίσης επισήμανε ότι υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για να αναχαιτιστεί η σεξουαλική βία στα κέντρα υποδοχή και διέλευση, που δεν εφαρμόζονται δυστυχώ. Δεν υπάρχουν ξεχωριστέ τουαλέτε για τι γυναίκε. Δεν έχουμε ξεχωριστού ε, χώρου ε, ε, διαμονή. Αισθάνονται ανασφάλεια οι γυναίκε και δεν λαμβάνονται υπόψη οι παγκόσμιε κατευθυντήριε γραμμέ. Επίση, χρειαζόμαστε περισσότερε εμπειρογνώμονε για τη σεξουαλική βία στα κέντρα αυτά. Επίση, να εξασφαλιστεί διερμηνία γιατί μερικές φορές όταν δεν καταλαβαίνουν ε, του ε, υπαλλήλου απευθύνονται στου λαθροδιακινητές γιατί δεν έχουν διερμηνέα για να τους βοηθήσει. Επίση, ε, θέλουμε και μηχανισμούς ενημέρωση συγκεκριμένων υποθέσεων άσκησης σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου. Αυτά μας είπε η κυρία Ρέιλι, πολύ σημαντικά και επισήμανε ότι η παρούσα πολιτική ασύλου δυστυχώς ε, θέτει σε κίνδυνο τις γυναίκες και χρειαζόμαστε κατεπηγόντως ε, κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ουτασούν και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα όσα μας μεταφέρατε από τις ομιλητές ε, πολύ σημαντικά για τα συμπεράσματά μας. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γιούτο που ήταν ε, η συγκήτρια στο δεύτερο εργαστήριο για την ε, υγειονομική περίθαλψη και την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των ετών των άσυλο. Κυρία Γιούτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σαφέστατα το εργαστήριο αυτό το οποίο παρακολούθησα είναι το πιο τεχνικό διότι αφορά τις πτυχές που αφορούν ε, την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται οι πρόσφυγες, κυρίως οι γυναίκες πρόσφυγες. Αυτό λοιπόν ήταν το ε, πλαίσιο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ε, έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη μετακίνηση μεταναστών και προσφύγων που φεύγουν από σειράξει, από διώξει ε, και πολλέ φορέ διώξει που βασίζονται στο φύλλο. Και οι, γυναίες, οι γυναίκες είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες κατηγορίες διότι βρίσκονται σε ικτρή κατάσταση στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Ιδίω αν πρόκειται για γυναίκες οι οποίες είναι μόνες, έγκυες, ε, που θυλάζουν στην εφηβεία και πολλό δε μάλλον το γεγονός ότι είναι γυναίκες που μπορεί να έχουν κάποια αναπηρία ή ε, μεγάλης Είναι σαφές λοιπόν ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις ε, και όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία τους πρέπει να είναι ε, πρωταρχικής φύσεως. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα και ε, ασχοληθήκαμε με διάφορα προβλήματα. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω ένα βήμα πίσω και να σας πω ποια είναι τα μέσα τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς ε, νομοθετικής. Υπάρχει οδηγία για την υποδοχή ε, των ε, όσων ζητούν διεθνή προστασία, οδηγία η οποία είναι ενισχύ, που λέει ότι οι ετούντε άσουλο έχουν δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και σε περίπτωση επίγουσα, αλλά και σε ειδικέ θεραπείε σε περίπτωση κάποια πάθηση. Επίση, ε, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγε έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβαση στην υγεία με τα υπηκόου των κρατών μελών. Και αυτό είναι κάτι σοβαρό γιατί δεν επαληθεύεται πάντα. Κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνε προβλέπονται επίση και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διακίνησης ε, ανθρώπων, ε, ψυχολογική συνδρομή, ε, συμβουλές και νομική συνδρομή όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για τη διακίνηση ανθρώπων. Επομένως η Ευρώπη διαθέτει τα νομοθετικά μέσα, αλλά υπάρχουν κάποιες επικρίσεις σε αυτή την περίπτωση. Ζητάμε να εφαρμοστούν όλα αυτά γιατί η οδηγία έχει μείνει τρόποντινά μόνο στα χαρτιά και δεν έχει υλοποιηθεί. Σήμερα το πρωί είχαμε και τα νέα στοιχεία της UNICEF του Φεβρουαρίου του 2016, επομένως πριν από λίγες ημέρες, όπου αναφέρεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 ο αριθμός των γυναικών και παιδιών που έφτασαν στην Ευρώπη ξεπέρασε κατά το διπλάσιο τον αριθμό των ανδρών και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η προσφυγική κρίση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά, τα παιδιά και οι γυναίκες είναι πλέον το 60% των προσφύγων και των ε, μεταναστών, ενώ τον Ιούνιο ήταν μόλις το 20%. Οι γυναίκες λοιπόν είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες ε, στον κίνδυνο βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης από τους διακινητές και από εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες συναντούν στη διάρκεια της διαδρομής τους. Ε, μας το υπενθύμησε και η Ναουάλ Σούφη. Ε, η Ευρώπη αρχίζει να γίνεται αδιαπέραστη. Δεν μπορούν να φτάσουν οι πρόσφυγες, αλλά είναι αδιαπέραστη και για το... Μάλλον είναι ιδιαίτερα διαπερατή στο οργανωμένο έγκλημα και τους ανθρώπους αυτούς που εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Αναφερθήκαμε επίση και στι δομέ και στι υπηρεσίε υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχει προσωπικό το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ενημερωμένο σε θέματα βία που βασίζονται ε, στο φύλλο και για να μπορέσουν να, παράξουν, να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη. Επίση πρέπει να υπάρξει ε, σύνδρομη προ το προσωπικό για να δίνονται πληροφορίε ε, στου ετούντε άσυλο και στου πρόσφυγε. Ένα από τα προβλήματα τα οποία ανέκυψε κατά τη συζήτηση είναι ότι υπάρχουν ελάχιστε μαρτυρίες γυναικών προσφύγων. Ε, ακούμε περισσότερο την άποψη των εθελοντών και του προσωπικού που ασχολείται με τους πρόσφυγες, αλλά έχουμε ελάχιστες άμεσες εμπειρίες, δηλαδή συνεντεύξεις ε, από γυναίκες πρόσφυγες και νομίζω ότι αναφέρθηκε και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και άμεσες εμπειρίες από ανήλικους, ασυνόδευτους ανήλικους που φτάνουν στην Ευρώπη, διότι υπάρχουν έφηβοι ε, που ε, είναι διαθέσιμοι, μπορεί να μιλήσει κανείς μαζί τους, μπορούν να υπάρξουν συνεντεύξεις αλλά και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς τους ασυνόδευτους ανηλίκους αυτή τη στιγμή. Τα κέντρα υποδοχής αυτή τη στιγμή έχουν πολύ ισχυρή ανδρική παρουσία, διότι υπάρχουν και ένοπλοι ε, και συνοριοφύλακες ε, και φύλακες εκεί και αυτό αποτελεί πρόβλημα για τις γυναίκες, διότι το γεγονός ότι είναι σχεδόν αποκλειστικά άνδρες και αστυνομικές δυνάμεις πολύ συχνά αποτελεί ανασταλτικό παράδειγμα και δημιουργεί προβλήματα και υπάρχουν και περιστατικά βίας. Καλό θα ήταν λοιπόν να αυξηθεί και ο αριθμός ε, των γυναικών μεταξύ του προσωπικού ασφαλείας που διαχειρίζεται τους πρόσφυγες. Όσον αφορά τις διαφορετικές πτυχές, ε, εδώ έχουμε την ανάγκη για να υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που να είναι καθαρά για γυναίκες και παιδιά. Να υπάρχουν χώροι στους οποίους να μπορούν να γίνουν εμπιστευτικές συνεντεύξεις στις οποίες αναφερθήκαμε πριν και για θύματα βίας, αλλά να υπάρχουν και ασφαλείς χώροι να αφήσει κάποιος τα παιδιά του ε, κατά την ε, θεραπεία, τους ελέγχους, παροχή θεραπευτικής αγωγής ή της συνεντεύξης. Επίσης πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη διανομή τροφίμων. Η Ναουάλ σήμερα το πρωί μας είπε ότι μπορεί να περιμένει κάποιος 3-4 ώρες ε, στο κρύο κάτω από τη βροχή για να πάει το καθημερινό του γεύμα. Αυτό ε, είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτο αν ε, αυτός ο οποίος περιμένει στην ουρά είναι μια γυναίκα έγκυος ή κάποιος ο οποίος έχει προβλήματα υγείας. Ε, και επίσης το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε νερό και σε ε, υγειονομικές εγκαταστάσεις. Επίσης, ε, αναφέρθηκε το πρόβλημα των ε, γυναικών εγγύων. Οι περισσότερε γυναίκε εγγύες έχουν και ε, σωματικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα και μπορεί να υπάρξει κίνδυνο θανάτου και της μητέρα και του βρέφου. Επομένω, πρέπει να παρέχονται κατάλληλε υπηρεσίε, οι οποίε πρέπει να θεωρούνται και ω ένα τρόπο, να παρέχουμε και άλλε υπηρεσίε. Πρέπει να μπορούμε να εξετάσουμε την κατάσταση τη υγείας όλων των γυναικών και να προβλέψουμε και μακροχρόνιε θεραπείε. Υπάρχουν όμω πάρα πολύ μεγάλοι φραγμοί στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχει δυσκολία επικοινωνίες, πολιτιστικέ πτυχέ, ε, ε, διαφορέ από, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υγεία και ακόμα και αν υπάρχουν γυναίκε οι οποίε ε, είναι πιο μορφωμένε και έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν κάποιε γλώσ, γλώσσε, μπορεί να μην γνωρίζουν από ιατρική, Επομένω, δεν μπορούν να περιγράψουν με κατάλληλού όρου τα συμπτώματά του και δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώ του συμβαίνει. Επίση, υπάρχει ανάγκη ανάγκη για ε, ε, θεραπευτική αγωγή και βοήθεια σε γυναίκες που είναι έγκυος ή σε ελεγχόνες ε, και υπάρχουν προβλήματα στη φροντίδα των παιδιών, δεν υπάρχει κατάλληλη συνοδός σε κάποιες περιπτώσεις. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν στη διάρκεια του εργαστηρίου είναι η κατεπίγουσα ανάγκη να ξεπεράσουμε όλους τους νομικούς ε, περιορισμούς που υπάρχουν για την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, κυρίως για τις γυναίκες εγγύους και για τα παιδιά. Πολλές γυναίκες οι οποίες, για παράδειγμα, θα πρέπει ε, κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο πρώτο κέντρο επιδοχής ε, να κάνουν και μία επίσκεψη σε γιατρό. Πολλές φορές οι γυναίκες αυτές αρνούνται να νοσηλευθούν γιατί υπάρχουν ε, άλλοι διοικητικοί και νομικοί φύσεως λόγοι. Μπορεί να φοβούνται είτε για οικονομικούς λόγους ή γιατί ε, φοβούνται να τις αναγνωρίσουν και μετά να τις ε, επαναπροωθήσουν αμέσως. Κάτι άλλο, αυτό αναφέρθηκε επίσης, η ανάγκη να παρέχεται ε, υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει υπόψη και την κινητικότητα. Δηλαδή να μην θεωρούμε μόνο ότι κάποιος μπορεί να έχει περίθαλψη σε ένα σταθερό σημείο σε μια χώρα, αλλά θα πρέπει ε, να παρέχεται και ε, φροντίδα σε περιοχές που σταθμεύουν αυτοί οι πρόσφυγες, παραδείγματος χάρη κινητές μονάδες που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν. Ε, είχαμε αρκετές οργανώσεις που συμμετείχαν, είχαμε μια εκπρόσωπο των γιατρών Χωρίς Σύνορα και ακούσαμε μια πολύ σημαντική μαρτυρία, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες οργανώσεις ε, που δραστηριοποιούνται, παραδείγματος χάρη Emergency, ε, που υποστηρίζουν και κυρίως βοηθούν σε λήψεις των κρατών μελών σε αυτές τις περιπτώσεις και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τους πάρα πολλούς εθελοντές όπως τη γυναίκα που υποδεχτήκαμε σήμερα το πρωί. Υπενθυμίζω την Ναουάλ Σαφ που είναι θελόντρια και έχει σώσει πάρα πολλέ ανθρώπινε ζωέ. Ε, οι αιτήσει ασύλου καθυστερούν πάρα πολύ για διάφορου διοικητικού λόγου. και αυτό φυσικά ε, σημαίνει ότι θα παραμείνουν και θα κρατηθούν περισσότερο στα κέντρα υποδοχή και αυτό μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τι γυναίκε. Ε, Κυρίω γυναίκε, οι οποίε ήταν αντικείμενο βία και κακοποίηση, Ε, ολοκληρώνοντας να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, εγγυηθούμε υγειονομική περίθαλψη σε όλε τι γυναίκε πρόσφυγε και ετούντε άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη. Έχουν διαφορετικέ απαιτήσει από του άνδρε, γιατί ορισμένε φορέ εκτίθενται σε πολλαπλού κινδύνους, ε, βία λόγω ε, φύλου, ε, επιπλοκέ κατά την εγκυμοσύνη και πολύ συγκεκριμένε θεραπευτικέ αγωγέ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένε φροντίδε, θεραπείε, οι οποίε παρέχονται βάση φύλου και πρέπει να διασφαλίσουμε ασφαλεί χώρου σε γυναίκε και παιδιά. Να υπάρχει φροντίδα και ε, ψυχολογική υποστήριξη για όλες αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά που υποφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, señora Σας ευχαριστούμε κυρία Αγιούτο. Τέλος, περνάμε στην τρίτη ομάδα εργασίας, στο τρίτο εργαστήριο, η κυρία Μπιόρκ. η η εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθήν Πέρτερ ε, και τους καλεσμένους που μίλησαν ε, στην ομάδα εργασίας μας. Είχαμε πολλές ε, μαρτυρίες από την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Τσεχία και άλλες χώρες επικεντρωθήκαμε στο θέμα της κοινωνικής ένταξης των γυναικών προσφύγων. Από τις μελέτες που ασχολήθηκα με το θέμα αυτό βλέπουμε ότι το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης είναι φλέγον. Και μάλιστα η ένταξη θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως. Δηλαδή ήδη από το ταξίδι. Η ένταξη ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο μας υποδέχεται η παγκόσμια κοινότητα στην πορεία προς τη χώρα προορισμού. Καλό θα είναι η εμπειρία αυτή του ταξιδιού να είναι θετική, για να δημιουργήσουν οι πρόσφυγες μια θετική εικόνα για την φιλοξενία που λαμβάνουν στα κέντρα υποδοχής και διέλευσης. Ε, κάποιοι συνάδελφοι μας μίλησαν ε, για τον παράγοντα χρόνο. Δεν θα πρέπει να χάνεται χρόνος ε, για την εκμάθηση μιας γλώσσας, ε, για την εκμάθηση ενός επαγγέλματος. Είναι σημαντικά στοιχεία της ένταξης. Επίσης, οι γυναίκες είναι το αγωνάρι της οικογένειας και η κοινωνική ένταξή τους θα κρίνει και την ένταξη ολόκληρης της οικογένειας στο νέο περιβάλλον. Μιλήσαμε και για διάφορα άλλα στοιχεία που άπτονται του κράτους πρόνοιας. Μιλήσαμε για τη σημασία που έχει η στέγη. Είναι σημαντικό να παρέχουμε στέγη ε, σε ένα κατάλληλο που να μπορεί ολόκληρη η οικογένεια να βρίσκει περίθαλψη, ώστε να μπορέσει πολύ πιο εύκολα να ενταχθεί κοινωνικά. Μιλήσαμε και για τη σημασία που έχει η εκμάθηση της γλώσσας. Επίσης, ε, να γίνεται αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων και πτυχίων από τη χώρα καταγωγής. Αλλά για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι σημαντική εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Οι γυναίκες πρόσφυγες ε, αντιμετωπίζουν πολύ συχνά ερωτισμό και προκαταλήψεις. Γι' αυτό θα πρέπει στις κοινότητας της υποδοχής ε, να καταπολεμήσουμε αυτές τις ρατσιστικές προκαταλήψεις, προκαταλήψεις που μερικές φορές ε, πλήττουν τις γυναίκες κυρίως. Επίσης μιλήσαμε για το μισθολογικό χάσμα. Υπάρχει διαφορά μισθολογική μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή η διαφορά είναι γνωστή και είναι αισθητή ακόμη και στις χώρες μας, αλλά είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό το μισθολογικό χάσμα ε, μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών γυναικών και οι γυναίκες πρόσφυγες ε, χρειάζονται έναν αξιοπρεπή μισθό, αξιοπρεπείς αμοιβέ που δεν θα είναι κατώτερες από τις αμοιβέ των ημεδαπών γυναικών. Θα πρέπει να λειτουργήσει το κράτος πρόνοιας ε, και αυτό υποθέτει ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και υποδοχή και φιλοξενία των παιδιών των γυναικών αυτών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Στο εργαστήριό μας μιλήσαμε και για τη σημασία που έχει η οικογενειακή επανένωση. Η οικογενειακή επανένωση φυσικά είναι κέριο στοιχείο της ε, κοινωνικής ένταξης. Γιατί αν ζει κανείς μακριά από την οικογένειά του, μακριά από τους ανθρώπους που αγαπά, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ενταχθεί στην κοινωνία της χώρας υποδοχής. Αυτό λοιπόν το σημείο θα πρέπει να μας απασχολήσει και σίγουρα τα παιδιά να μεγαλώνουν στις οικογένειές τους, να μην υποχρεώνεται κανένα παιδί να μεγαλώνει μακριά από τους γονείς του, μακριά από την οικογένειά του. Επίσης μιλήσαμε για τα εθνικά συστήματα υγείας. Βέβαια αυτό το ζήτημα απασχόλησε και το δεύτερο εργαστήριο. Μιλήσαμε και για το θέμα της ασφάλειας και της προστασίας. Δεν θα πρέπει οι γυναίκες πρόσφυγες στις χώρες υποδοχής να είναι και πάλι εκτεθειμένες σε ανασφάλεια. Γιατί και πάλι εκτίθενται στον κίνδυνο της ανασφάλειας ε, και δεν ε, νιώθουν ασφαλείς στη χώρα υποδοχής, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ενταχθούν στην κοινωνία. Γιατί αν υπήρχονται δεύτερη φορά επιθέσεις ε, από τις αστυνομικές δυνάμεις ή από τους διάφορους φορείς της χώρας υποδοχής, είναι σαν να βιώνουν το τραύμα δεύτερη φορά, κάτι που επιβραδύνει φυσικά πολύ περισσότερο την κοινωνική του ένταξη. Στην πράξη έχουμε πολλές ε, καλές πρωτοβουλίες ε, και από εθελοντικές οργανώσεις και από την κοινωνία των πολιτών και μάλιστα χάρη στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Ε, Αναβάνουμε γνώση των πραγματικών αναγκών. Και κρίμα είναι που πολλές φορές δεν ακούμε αρκετά τις εκκλήσεις που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η δικαστική συνδρομή, η νομική αρρωγή. Αν δεν γνωρίζει κανείς τα δικαιώματά του και τι κατοχυρώνεται από τον νόμο, είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί κοινωνικά ή να διεκδικήσει μια επαγγελματική κατάρτιση. Και το νομικό λοιπόν ζήτημα, η νομική πτυχή είναι πολύ σημαντική. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι στην έκθεση της ε, του τρίτου εργαστηρίου, μιλήσαμε και για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους πρόνοιας και τη σπουδαιότητα της οικογενειακής επανένωσης, που δυστυχώς δεν γίνεται σεβαστή σε πολλές χώρες, ακόμη και στη δική μου πατρίδα, τη Σουηδία. Είναι σημαντικό να τεθεί ένα τέρμα στη διακριτική μεταχείριση και στις προκαταλήψεις ε, που μαστίζουν κυρίως τις γυναίκες. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα του τρίτου εργαστηρίου και ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό. Muchas gracias, señora Björk. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπιόρκ. Μια και ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των συμπερασμάτων των τριών εργαστηρίων, μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Ήδη έχουμε συντάξει ένα κατάλογο με ομιλητές. Αν επιθυμεί και άλλος το λόγο, παρακαλώ να το δηλώσει για να τον εγγράψουμε στον κατάλογο. Μπορείτε να συμπληρώσετε ε, τα στοιχεία σας και να το δώσετε στη γραμματεία για να σας συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των αγορητών. Τρία λεπτό καθένας παρακαλώ. Ξεκινάμε με την κυρία Σεσίλ Κέγκε, που είναι ευρωβουλευτής και η εισηγήτρια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ. Αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητές φίλες, αγαπητές αδελφές μου. Είναι χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να μιλώ και πάλι εδώ στην Ολομέλεια ε, και μάλιστα επί τη ευκαιρία ε, του εορτασμού της ημέρας της γυναίκες. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο ε, αναφανδόν υπέρ είμαι υπέρ της άρσης οποιασδήποτε μορφής ε, διάκρισης. Ε, η βοήθεια προς τους πρόσφυγες σημαίνει καταρχάς διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ε, ε, χιλιάδων και εκατομμυρίων γυναικών, κοριτσιών και παιδιών που έρχονται στα κράτη-μέλη μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των γυναικών που φεύγουν δεν καταφέρνουν να ζητήσουν άσυλο στο εξωτερικό. Η πορεία τους σταματάει πολύ νωρίτερα. Αυτές που τα καταφέρνουν όμως ε, δεν σημαίνει ότι ε, φτάνουν πάντα στη σωτηρία. Δεν είναι πάντα το άθλο συνώνυμο της σωτηρίας. Ε, στις χώρες προορισμού ή στις χώρες διέλευσης υπάρχουν πολύ σοβαρά περιστατικά βίας όπως γίνεται και στην χώρα που θα τους υποδεχθεί. Οι γυναίκες που ζητούν άτεσιλο χρειάζονται πολύ συγκεκριμένη προστασία και είναι τελείως διαφορετική από αυτή των ανδρών. Και στο πρώτο στάδιο της υποδοχής όπου θα πρέπει να τους εγγυηθούν όχι μόνο κατάλληλοι στέγη και ε, υπηρεσίες αλλά και ψυχολογική υποστήριξη μέσω της ε, σχετικά άγνωστης ψυχής, ε, πτυχής της εθνοψυχιατρικής, η οποία λαμβάνει υπόψη και την καταγωγή του ανθρώπου και τις απαιτήσει λόγω της ε, διαφορετικής νοοτροπίας που υπάρχει στην ογειονομική περίθαλψη. Και κυρίως πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη μεταχείριση και την κράτηση γυναικών και παιδιών και κατά το πρώτο στάδιο της υποδοχής, όπου θα μπορεί να υπάρχει συνδρομή από γυναίκες και στο στάδιο της ε, κοινωνικής ένταξης ε, ε, για τη βοήθεια στην παιδεία και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης, είναι το μέλλον του κόσμου. Η έκθεση της ε, Mary Hannibal, η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών στην έκθεση πρωτοβουλίας, ε, στην οποία είμαι συνεισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, ε, η ίδια η έκθεση πρωτοβουλίας αποτελούν το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να εκπονηθεί μια μεταναστευτική πολιτική, η οποία θα συνάδει με τις θεμελιώδεις αξίες μας θα κάνω την ίδια έκκληση που έκανε και η Μέρι Ρόμπινσον. Εμείς γυναίκες ε, πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να εισακουστεί η φωνή μας στα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια κυρίως τις 7 18 και 18 ε, και 19 Μαρτίου. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να αντιταχθούμε στις μειοπικές και εγωιστικές πολιτικές ε, του περιορισμού των προσφύγων, του κλεισίματος των συνόρων και, της, ε, ε, και του περιορισμού της νόμιμης μετανάστευσης. Το μεταναστευτικό πρέπει να το διαχειριστούμε, όχι να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κατάστροφη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων και επίσης θα πρέπει να το διαχειριστούμε διαχειριστούμε εγγυόμενοι ε, νόμιμες και ασφαλείς οδούς ε, μετανάστευσης, δημιουργώντας ε, κανάλια μόνιμης μετανάστευσης και εντάσσοντας τους μετανάστες στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό ιστό των χωρών μας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με το ίδιο μήνυμα ελπίδα ε, που ε, μας έδωσε και η Ναουάλ Σουφή. Μόνο με ενωμένε τι δυνάμεις μας και μόνο ε, να εισακουστεί η φωνή μα, θα μπορέσουμε να ξαναδώσουμε στη Μεσόγειο το πραγματικό της χρώμα, το γαλάζιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκλησή σα. Είμαι στη διάθεσή σα να δώσω μάχη μαζί σα. Ευχαριστώ πολύ. Eh, ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Κιέγγε. Τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Φεντερίκα από Φεντερίκα από την Βουλή της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το ζήτημα. Συζητάτε πολύ στην Ιταλία που, ε, ε, από την οποία κατάγομαι. Η Ιταλία λόγω γεωγραφικής της θέσης είναι πιο εκτεθειμένη από άλλες χώρες. Είμαστε εκτεθειμένοι μόνιμα στο μεταναστευτικό μέσο θαλάσσης. Και φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα και υπάρχουν και προφανείς περιορισμοί. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών κυρίως και των ανηλίκων, δηλαδή των πιο ευάλωτων ομάδων μεταναστών δυστυχώς η Ευρώπη δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσει και τα αίτια αυτού του φαινομένου, οικονομικά, πολιτικά και αίτια αλλά και ε, λόγω πολέμου. Ε, μόνο αντιμετωπίζοντας αυτά τα αίτια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες και να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές ροές. Θα ήθελα να σταθώ εντάχει σε δύο ουσιώδη θέματα τα οποία συζητήθηκαν ε, ίσως ε, και λίγο πιο ε, εκτενός από την κυρία Σούφη, η οποία αναφέρθηκε σε μαφία. Μαφία η οποία δυστυχώς ε, διαχειρίζεται σχεδόν αποκλειστικά την κίνηση και την εμπορία των μεταναστών, κυρίως στη χώρα μου, στην οποία δεν υπάρχουν ανθρωπιστικοί διάβλοι νόμοι μεσοδοί οι οποίε θα ήταν απαραίτητε για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και να μην υπάρχει εκμετάλλευση από πλευράς οργανωμένου εγκλήματο. Επίση, θα ήθελα να επιστήσω και την προσοχή όλων σα ε, και στην ανάγκη να υπάρχει μια μόνιμη χρηματοδότηση εντός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι σε όλες τις χώρες ε, θα υπάρχει υγειονομική, ψυχολογική περίθαλψη, κατάλληλη ε, βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη και το πόσο ευάλωτοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι από αυτή τη συζήτηση να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει και μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. από την Επιτροπή Γυναικών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Σόντρο. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στην Τσεχική. Ναι, και είναι και πιο εύκολο για μένα. Κυρίε και κύριοι. Ξέρω ότι είναι προσκεκλημένοι. Με μεγάλη χαρά δράτω με τις ευκαιρίες να σας απευθύνω το λόγο εκ μέρους ε, των συναδέλφων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στερόμεθα ευγνώμονες για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για τα θέματα αυτά. Είναι πολύ, σημερινή, πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Μια ημέρα που αναγνωρίζεται ο ρόλος της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, θα θέλαμε να πάρουμε και εμείς τις σκητάλη στα χέρια μας για την επόμενη, για την εκδήλωση της επόμενης χρονιάς. Οι γυναίκες μετανάστες αντιμετωπίζουν διτές δυσκολίες. Όχι μόνο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της Ευρώπης χαμηλότερους μισθούς, τον κίνδυνο τη βία κτλ. Οι μετανάστριες όμως έχουν ε, να αντιμετωπίσουν και την ξενοφοβία. Τις βλέπουν σαν ξένες, σαν ολοδαπές. Και γι' αυτό πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε στέγη, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, υποστήριξη στα θύματα της βίας, υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν μικρά παιδιά να φροντίσουν. Γιατί αυτά συνήθως δεν προλαβαίνουν να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Πρέπει να στηρίξουμε γυναίκες κορίτσια, μικρά παιδιά. Ξέρετε ότι 10.000 μη συνοδευόμενα ανήλικα παιδιά βρίσκονται στην Ευρώπη, εκτεθειμένα να πάσα στιγμή στο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε επιτύχει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και ιδιαίτερα θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη δουλειά που κάνουν οι φιλανθρωπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να γνωριστεί η δουλειά των εθελοντών. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να αναγνωρίσουμε το ρόλο, την προσφορά των εθελοντών. Πρέπει να στραφούμε προς αυτούς, να πάμε να τους μιλήσουμε, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν από την εμπειρία του. Αλλά πρέπει να είμαστε και 28 διαφορετικές χώρες στην Ένωση αναζητούν μια κοινή προσέγγιση με διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο όμως, με διαφορετικές εμπειρίες. Εμείς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια, χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να προσεγγίσουν το θέμα με γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προστασία της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής. Πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να παρεμβαίνουμε. Και κάτι που δεν έχει ακουστεί πιστεύω αρκετά. Η λύση για όλα αυτά είναι η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Η νύχηση ασφάλειας στις Αφρικανικές χώρες και τη Μέση Ανατολή, η υποστήριξη Οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Γιατί αν είναι ασφαλείς οι άνθρωποι στις χώρες τους, αν βρίσκουν δουλειά στις πατρίδες τους, δεν θα χρειαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους. Και αυτό ισχύει για όλες τις γυναίκες για τις οποίες μιλήσαμε, για όλα τα παιδιά και για όλες τις οικογένειες. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν ε, συνυπευθυνότητα, ισχύει αρχή της επικουρικότητας και γι' αυτό ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τα όσα έχουν αναλάβει ως ευθύνη, το δικό τους μερίδιο. Αλλά μόνο από κοινού μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη να φέρει αποτελέσματα. Και η γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο είναι ότι οι γυναίκε και τα παιδιά πρέπει να πάνε πρώτα, να προστατευτούν κατά προτεραιότητα. Σα ευχαριστούμε κυρία ε, Σόιντροβα, η κυρία Σδεμίρα από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. ξέρετε, κυρίε και κύριοι συναδελφοί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών οργανώνεται αυτή τη συνεδρία. και θέλω να σα ευχαριστήσω για την ε, πολύ σημαντική αυτή πλατφόρμα. Η Επιτροπή το τουρκικό κοινοβούλιο έχει την Επιτροπή Ισότητα Ευκαιριών για τις γυναίκε και του άντρες. Είμαστε μέλη αυτή και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και ταυτόχρονα να τονίσουμε την αυτοθυσία με την οποία η χώρα μας υποδέχεται τους πρόσφυγες στην ε, Τουρκία. Η Φίλιος είναι μάρτυρας ε, της μεγαλύτερης εξόδου προσφύγων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε να κάνουμε με συνεδρίαση σήμερα στην οποία εντατικά συζητούνται όλα αυτά τα θέματα των προσφύγων γυναικών και οι ανάγκες για την παροχή προστασία σε αυτές. Η τελευταία πενταετία έχει φέρει με την εκκίνηση του πολέμου στη Συρία στην Τουρκία πολλούς πρόσφυγες. Έχουμε 900 χιλιόμετρα σύνορα χερσαία με τη Συρία και πάρα πολλούς πρόσφυγες που έχουν περάσει το ίμιση δε αυτών των προσφύγων είναι γυναίκες. Πολύ μεγάλο ποσοστό μικρά παιδιά. Η Τουρκία έχει διατηρήσει πολιτική ανοιχτών συνόρων όλα αυτά τα χρόνια και έχει σταθεί πραγματικό σύμμαχος στην γείτονα Συρία. Έχουμε περί τα 3 εκατομμύρια Σύρων προσφύγων στην Τουρκία εκ των οποίων ε, το 50% περίπου είναι σε πολύ νεαρή ηλικία και το 50% επίσης γυναίκες, είπε η κορίτσια. Έχουμε περίπου 200.000 ε, πρόσφυγες από τη Συρία σε καταπλησμούς. Έχουμε δαπανίσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ε, περίθαλψή τους και εγώ ως εκπρόσωπος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ήθελα να σας πω ότι το πρόβλημα αυτό των προσφύγων στη Συρία δεν το προσφύγων από τη Συρία που βρίσκονται στην Τουρκία δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί μόνη της η χώρα μας να επιλύσει. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως τα κράτη-μέλη αυτής να δείξουν αλληλεγγύη προς Τουρκία και να προσφέρουν υποστήριξη ανεπιφύλακτη σε κάθε διάσταση του προβλήματος των προσφύγων και ιδιαίτερα η χώρα μας που έχει και στρατηγική σημασία εν ώψη του προσφυγικού αυτού προβλήματος πρέπει να στηριχθεί ταχύτατα και οικονομικά για να αναπτύξει τις δομές υποδοχής των προσφύγων. Τα προβλήματα είναι γνωστά, είναι ξεκάθαρα, τα εξέθεσαν οι πάντε εδώ και πρέπει κατεπηγόντω να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να αναλυθεί δράση κατεπηγόντω. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, πρέπει να διατεθούν το ταχύτερο δυνατό τα κονδύλια που χρειάζονται για να υλοποιηθούν τα προγράμματα, για να εφαρμοστούν τα μέτρα και πρέπει με το προενταξιακό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατεθούν το ταχύτερο δυνατό κονδύλια για να υποστηριχθεί η Τουρκία. Ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές της χώρας μας έχουμε αντιμετωπίσει ε, με ένταση προβλήματα σχετικά με τους πρόσφυγες. Εμείς ως αντιπολίτες εξωματική υποστηρίζουμε την κυβέρνηση μας σε όλες τις προσπάθειες για την μετώπιση των προβλημάτων που γεννούνται από το προσφυγικό, από την προσφυγική κρίση. Πάνω απ' όλα βεβαίως θέλουμε να σταματήσει ο εμφύλιος πόλεμος στην Συρία, ο οποίος είναι και η κύρια πηγή για την έξοδο από τη χώρα τους αυτών των προσφύγων, κυρίως γυναίκων και παιδιών, πρέπει όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουν καταφύγιο ασφαλές στους ανθρώπους αυτούς και να βοηθήσουν να σταματήσει ο πόλεμος. Ο ιδρυτής του ε, ιστορικού μας κόμματος, ο Μουσταφά Μάλατα Τατούρκο, είχε ε, πει μια ιστορική φράση «Ειρήνη στη χώρα μας, ειρήνη στην πατρίδα μας, αλλά και ειρήνη στον κόσμο». Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο κινούμαστε, ειρήνη στην ε, χώρα μας, αλλά και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Οι πρόσφυγες από τη Συρία που ζουν στη χώρα μας, έχουν ανάγκη και από συνθήκες οικονομικές, κοινωνικές, ε, εκπαιδευτικές, ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαψης και άλλες τις οποίες ε, διαθέτει η χώρα μας και εμείς από τη Βουλή τους υποστηρίζουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πρέπει ωστόσο να βρεθούν και λύσεις σχετικές με το νομικό καθεστώς των προσφύγων. Εμείς είμαστε συμβαλόμενο κράτος στη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Προσφέρουμε στο βαθμό που μπορούμε την υποστήριξή μας και την προστασία μας, αλλά είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές μας και για λόγους γεωγραφικούς. Με τις ρυθμίσεις που έχουν περάσει από την ε, Βουλή, η Μεγάλη Τουρκική συνοσυνέλευση. χορηγήσαμε το 2014 το καθεστώς προσωρινής προστασίας σε όλους τους Σύρους, που τους επιτρέπει και να έχουν κοινωνική ε, πρόνοια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση κτλ και βέβαια δυνατότητα απασχόληση στη χώρα μας. Κλείνοντας θα ήθελα να πω, ζητώντα συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο μου, το χρόνο μου ότι πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και στην αντιμετώπιση του προσφυγικού αλλά και στην, στην ένωση με την Τουρκία. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία ε, είναι χαρακτηριστικά της ιστορίας μας, δείχνουν μεγάλους, ε, μεγάλα δεινά και ταλαιπωρία. Ε, λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά ήδη σας δώσαμε διπλάσιο χρόνο από όσο δικαιούσασταν. Είχαμε πει τρία λεπτά, Ήδη μιλάτε έξι λεπτά. Σας είχαμε παρακαλέσει να περιοριστείτε στο τρίλεπτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απόλυτη συνείδηση της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία και φυσικά είναι απαραίτητη η συνεργασία με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Μάλιστα πριν από ένα χρόνο στην αντίστοιχη εκδήλωση με θέμα τις γυναίκες και την παιδεία, μία συνάδελφός σας από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση μας είχε προειδοποιήσει για αυτό που συνέβαινε και Ήδη ένα χρόνο μετά είδαμε ότι τελικά όλα αυτά που μας προειδοποιούσαν, για τα οποία μας προειδοποιούσαν, έγιναν πραγματικότητα. Και φυσικά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε να μονοπολείτε το χρόνο αγόρευσης. Από την Γερμανική Βουλή τώρα, η κυρία και Χίλε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ ως μέλος ε, του τοπικού Κοινοβουλίου του κρατηδίου της Βρέμης. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία αυτή και βέβαια για την πολύ σημαντική έκθεση η οποία εκπονείται εδώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις για την έκθεση και ξεκινώ με το πρώτο σημείο που είναι βέβαια οι λόγοι της φυγής, οι λόγοι της προσφυγιάς που πολλοί συνάδελφοι εξέθεσαν νωρίτερα. Δύο είναι σημαντικοί λόγοι τα γίνουν έτσι αυτής της ε, ακραίας κατάστασης, της φυγής, της προσφυγιάς, της αίτηση για το άσυλο, για όλες τις γυναίκες και όλους τους πρόσφυγες, όχι μόνο αυτούς που έρχονται στην Ευρώπη, αλλά τα 60 εκατομμύρια ανά τον κόσμο που βρίσκονται στο δρόμο της προσφυγιάς και αυτό, αυτά τα γενουσιοργά αίτια είναι ο πόλεμος. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε ε, ξεκάθαρα. Είναι άλλωστε μια από τις παλαιότερες διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος της Ευρώπης ε, η ε, κατάπαυση των πολέμων. Η Συρία βρίσκεται τώρα σε έκτο χρόνο εμφύλιου πολέμου. Πρέπει και εμείς ως γυναίκες να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα, αποστέλουμε την ειρήνη. Το άλλο θέμα βέβαια είναι η πείνα. Ο άλλος λόγος είναι η πείνα. Και εδώ στις Βρυξέλλες, από τις Βρυξέλλες θέλω να πω ότι η γεωργική πολιτική εξακολουθεί να έχει σαν συνέπεια την ε, ε, ανάδειξη λιμών και καταστάσεων προβληματικών σε διάφορες περιοχές του κόσμου που οδηγούν τις γυναίκες και τα παιδιά τους να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Κάτι ακόμη. Στο σημείο 18 της εκθέσεως, η αναφορά σε χώρες ασφαλής προελεύσεως. Είναι καλό το ότι αναφέρεται αυτό στην έκθεση. Δεν πρέπει με τα όσα συζητούνται και στη Γερμανία εντατικά η ανάδειξη ασφαλών χωρών προελεύσεως να σημάνει ανέρεση του δικαιώματος στο ε, άσυλο. Για άλλη μια φορά νομίζω και πρέπει να το επαναλάβουμε, πάντοτε πρέπει να επαληθεύεται αν υπάρχουν σε συγκεκριμένη περίπτωση, ανεξάρτητος του αν κάποιος πρόκειται από ασφαλή, ως ασφαλή χαρακτηριζόμενη χώρα, ε, δικαίωμα στο άσυλο για συγκεκριμένου λόγους. Και επίσης δεν βλέπω στην έκθεση πουθενά αναφορά σε προγράμματα επανεγκατάστασης. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καλύτερη λύση και για τις γυναίκε μέσω του ε, τι είπα τι αρμοστές των ΗΠΑ για του πρόσφυγες να έχουν τη δυνατότητα για την επανεγκατάσταση έτσι ώστε όλη αυτή η δύσκολη διαδικασία της φυγής και της προσφυγιάς, η έκθεση ε, στην εκμετάλλευση της μαφίας και των λαθροδιακινητών να προχωρούσε πιο απρόσκοπτα. Πρέπει να υποστηρίξουμε προγράμματα επανεγκατάσταση. Υπάρχει άλλωστε μια οδηγία ευρωπαϊκή για υποδοχή ε, προσφύγων δεν έχει όμως ακόμη προχωρήσει σε εφαρμογή. Αυτό θα έχει βέβαια σε συνέπεια και μεγάλο κόστος και εξοικονόμηση κόστους δαπανών αλλά οπωσδήποτε και απαλλαγή αυτών των γυναικών και των παιδιών τους από πολλά δεινά εάν μπορούσαν κατευθείαν από το Λίβανο, από την Ιορδανία ή από άλλα κράτη τα οποία βρίσκονται να γίνονται δεκτά, δεκτές κατευθείαν για επανεγκατάσταση. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την έκθεση. Χαίρομαι για το γεγονός ότι γίνεται παραπομπή και στα Ηνωμένα Έθνη στο σημείο 5 της εκθέσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ε, Ευρώπη να διατηρήσει την προσήλωσή της αυτές τις αρχές. Μας έχουν απομείνει μόνο 10 λεπτά για τη συζήτηση. Ως εκ τούτου, θέλουμε παρακαλώ τους επόμενους ομιλητές, τις επόμενες ομιλήτριες να είναι όσο πιο λακωνικές γίνεται για να μιλήσουν όσο περισσότεροι συνάδελφοι μπορούν. Αλλιώς θα πρέπει να διακόπτω δυστυχώς. Η κυρία Άιρα Κορόμπικ από τη Σερβική Βουλή. Η κυρία Άιρα Κορόμπιτς από τη Σερβική Βουλή. Τσόροβιτς. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω σερβικά. Δεν πρόκειται να σας διαβάσω αυτά που έγραψα ήδη από το Βελιγράδι, γιατί μετά από την συζήτηση έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι ρητορική. Όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Αρκούν λοιπόν τριάμιση μόνο ώρες για τη συζήτηση αυτού του τόσο σημαντικού ε, θέματος. Φυσικά ε, είναι κοινή ευθύνη να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και να αναλάβουμε και συγκεκριμένες ε, δράσεις. Γι' αυτό θα ήθελα τους επόμενους μήνες αυτό το θέμα να παραμείνει στο επίκεντρο, στο επίκεντρο της συζήτησης. Όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα. Η δεύτερη ερώτηση δεν είναι ρητορική, είναι η ερώτηση επί της ουσίας. Φυσικά μιλήσαμε σήμερα για τους πρόσφυγες, πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ, αλλά δεν είχαμε προσκαλέσει ούτε μία γυναίκα από τι χώρες αυτές. Για μένα το καλύτερο που άκουσα ήταν η εμπειρία των γυναικών της εθελόντριας που είχε επιτόπου έργο. Καλό θα ήταν όμως να, να ακούσουμε τις μαρτυρίες από τις ίδιες τις γυναίκες. Νομίζω είναι σύγκριτη δική τους εμπειρία και τα δικά τους βιώματα θα πρέπει να ακούσουμε. Η τρίτη ερώτηση είναι υποθετικού χαρακτήρα και δεν περιμένω καν απάντηση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα κάθε ένας από εμά να βάλει το χέρι στην καρδιά και να πει, αν κάποιο σήμερα μας ε, πει ε, ε, ότι έχετε ε, την επόμενη εβδομάδα ένα λεωφορείο από τις Βρυξέλλες για να περάσουμε τρεις-τέσσερις εβδομάδες σε ένα καταβλισμό προσφύγων. Θα θυσιάζαμε τον πολύτιμο χρόνο μας για να περάσουμε τρεις-τέσσερις εβδομάδες σε, μια, σε ένα καταβλισμό προσφύγων με ψυχολογική υποστήριξη, με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ερωτώ λοιπόν και απαντήστε με το χέρι στη καρδιά. Υπάρχει κάποιο από εμά που θα ήταν έτοιμο να πάει τρει-τέσσερι εβδομάδε σε ένα καταβλισμό προσφύγων και να μείνει μαζί με του πρόσφυγε για να δει τι περνάνε. Ευχαριστώ. Στο Ισαγουρά Είμαι βέβαιη πω ναι. Έχει το λόγο η κυρία Μαπρονικόλα από το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να πω ότι, όπως είπα και προηγουμένως στο workshop, για μας το προσφυγικό ζήτημα στην Κύπρο δεν προσεγγίζεται φιλοσοφικά, ακαδημαϊκά, πολιτικά και ιδεολογικά μόνο. Εμείς έχουμε βιώσει την προσφυγιά ως Κύπροι και την βιώνουμε εδώ και 40 χρόνια. Τα συναισθήματα, πιστεύστε με, είναι τα ίδια και εγώ συμφωνώ με την προηγούμενη συνάδελφο ότι έπρεπε να έχουμε εδώ πρόσφυγες από τη Συρία, από το Ιράκ, για να μας πούν τα συναισθήματα τους. Γιατί τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων είναι τραγικά. Χάνουν την ταυτότητα τους, χάνουν την αξιοπρέπεια τους, προσπαθούν να, να δώσουν φαΐ και ασφάλεια στα παιδιά τους, πεθαίνουν καθημερινά στη θάλασσα της Μεσογείου και είναι τραγικές οι συνθήκες που βιώνουν στα ελληνικά νησιά οι εθελοντές ε, στη Λέσβο, στην ΚΟ και είναι και σε αυτούς που πρέπει να δώσουμε ένα χέρι στήριξης και υποστήριξης θα πρέπει να δώσουμε όχι μόνο οικονομική βοήθεια αλλά να δώσουμε και χέρι ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλο το τίμημα που πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι για να προχωρήσουν προς την ελευθερία, έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε ανοιχτά τα σύνορα, έχουμε υποχρέωση να τους δώσουμε αξιοπρέπεια και να επανεγκατασταθούν μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους και τελειώνω λέγοντας ότι οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι 60 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες σε όλον τον κόσμο. 20 εκατομμύρια έχουν διαφύγει σε άλλες χώρες, 18 εκατομμύρια παραμένουν στις χώρες τους εκτοπισμένοι. 4 εκατομμύρια βρίσκονται στο σπίτι μας, στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη η αριθμοί και είναι και πολύ μεγάλες οι δικές μας οι ευθύνες. Πρέπει να βοηθήσουμε πρακτικά. Ευχαριστώ για Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και εντός των χρονικών ορίων. Να πω και στην προηγούμενη ομιλήτρια ότι στο πρώτο εργαστήριο ε, είχαμε μία πρόσφυγα από το Ιράκ θα μπορούσαμε βεβαίως να είχαμε καλέσει περισσότερους ακτιβιστές ε, και ανθρώπους ε, ε, πρόσφυγες, αλλά να σας πω ότι δώσαμε το λόγο σε μια πρόσφυγα σε ένα από τα εργαστήρια. Να δώσω τώρα το λόγο στη Σουζάνα Μαντόρα από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη διοργάνωση της εκδήλωσης για ένα τόσο σημαντικό θέμα, ένα θέμα, ένα θέμα ζωτικής σημασίας που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών ε, προσφύγων και του ανάσυλων. Ε, είχαμε μια πολύ σημαντική έκθεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια πρόοδο σε αυτό το θέμα ε, της δίωξης των γυναικών και της βίας λόγω και το νομικό και το ουσιαστικό ζήτημα θα πρέπει ε, της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνία ολίθο κάθε κοινωνία. Σχεδόν σε όλες τις ε, κοινωνίες και σε όλους του τομείς δραστηριοτήτων οι γυναίκες είναι θύματα ε, ανισοτήτων και de facto και de jure ανισοτήτων. Και παρόλο που οι συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλες τις χώρες, οι διακρίσει εις βάρος των γυναικών διονύζονται εξαιτία τη ύπαρξη στερεοτύπων, ε, πρακτικών και θρησκευτικών ή πολιτιστικών παραδόσεων που είναι εις βάρος των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να, να ε, λάβουμε υπόψη τη θέση των γυναικών υπό τη σκοπιά του φίλου και να πατάξουμε οποιαδήποτε βιαιότητα εις βάρος των γυναικών. Επίσης θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν την ε, προέλευση, διέλευση, ε, καταγωγή ε, και προορισμό και τις συνθήκες που συνοδεύουν όλο αυτό το ταξίδι. Επίσης, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες πρόσφυγες στην παιδεία, να εξασφαλιστεί η διαβίου κατάρτιση και η δική τους αλλά και του διδακτικού προσωπικού με, ιδιαίτερο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε την Σύμβαση της Γενέβης του 1951 ε, που αναφέρει ήδη ότι οι γυναίκες θύματα ε, συμπεριφορών ε, εξαστηλιστικών για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που έχουν φιλετικό χαρακτήρα φύλου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στην Πορτογαλία έχουμε διώξει των γυναικών λόγω φύλου και δυστυχώς ε, ε, τη μόνο μόνο κουρική προστασίας. Δεν είναι ε, το ίδιο με την προστασία που κατοχυρώνει η Σύμβαση της Γενέβης στο αρθρο 1α. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία για βίες βάρος των γυναικών και να διαδώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Και ιδιαίτερα στις χώρες υποδοχής αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να θεωρηθούν ως ασφαλής νέα αρχή για τη γυναίκα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα από την κρατική νομοθεσία και να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερα στι ε, επεξεργασίε των αιτήσεων αλλήλου. Βέβαια, άλλο ο νόμο και άλλο η έμπρακτη εφαρμογή του νόμου, που στην περίπτωση τη Πορτογαλία δυστυχώ ε, υπάρχει μεγάλη ακόμη απόσταση. Επίση, θα πρέπει να γίνει μια διαπαιδαγώγηση και των μέσων μαζική ενημέρωση, ε, που είναι σημείο κλειδί στο, στο όλο αυτό θέμα. Γιατί η πραγματική αλλαγή της νοοτροπίας θα πρέπει να ξεκινήσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη γυναικεία παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, για να γίνει πιο ε, εμβρηθή ανάλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Να αφήσουμε την επιφανειακή προσέγγιση. Θα πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί ε, γιατί μόνο έτσι θα πατάξουμε τις προκαταλήψεις. Και περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Ε, χρειαζόμαστε το Σέγγεν και επαναφορά στις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης ε, του ονείρου που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύει τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Ευρώπη είναι τα θεσμικά της όργανα. Και ένα από αυτά που εκπροσωπούνται τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα πρέπει να αναλυθεί η δέσμευση της ε, τήρησης των ηλυμένων υποχρεώσεων. Η κυρία Σλάμπεριγουάν από την Αυστριακή Βουλή, παρακαλώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Τα ίδια πάλι. Τα κράτη τα οποία απέστρεφαν το βλέμμα όταν εκδηλώνονταν ο πόλεμος, τώρα είναι αυτά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν τις ροές των προσφύγων. Και πολλά είναι τα κράτη που λένε «Α, είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα προβλήματα της κρίσης, Αλλά για την ουσία δεν μιλάει κανείς. Εκεί λοιπόν ακριβώ, εδώ που είναι τόσες πολλές οι γυναίκες μέσα σε μια συνεδρίαση, συνεδρίαση είναι νομίζω η ώρα να μιλήσουμε για την κατάσταση και των γυναικών στις χώρες μας, των πολιτικών, που θέλω να σας υπενθυμίσω, των γυναικών που έχουν βιάσει τα μέλη του Ισλαμικού κράτους, που τις έχουν πουλήσει σκλάβες, που έχουν κινηθεί από δίκτυα και που ακόμα δεν έχουν ε, βρεθεί. Μόνο ένας μαζικός τάφος γυναικών βρέθηκε πριν από μερικούς μήνες, αλλά η διεθνής κοινότητα δεν κούνησε ούτε το μικρό της δαχτυλάκι όπως και τα κορίτσια που είχαν απαγάγει από την Μπόκο Χαράμ, οι τρομοκράτες, για τα οποία είπανε «Α, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτά μεγαλώσαν, έχουν μείνει και έγκυοι, έχουν κάνει και παιδιά, τι να κάνουμε τώρα εμείς». Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τουλάχιστον την ευθύνη αναζήτησης των θυμάτων και αποκατάστασης της αξιοπρέπειάς τους, μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και πάλι και για τους ανθρώπους αυτούς που φτάνουν στις χώρες μας, πάλι δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να, ε, ακούσαμε από την Τουρκία ότι έχουμε τόσους πολλούς πρόσφυγες πάρει, είμαστε σε κατάσταση απελπισίας, χρειάζεται να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είπε κανείς όμως ότι στην Τουρκία είναι πολλές οι γυναίκες πρόσφυγες οι οποίες πέφτουν θύματα μαζικού εμπορίου ανθρώπων που τις πουλάνε και τις αγοράζουν, που τις δίνουν σε καταναγκαστικούς γάμους, που προσπαθούν και αγωνίζονται μόνο για την επιβίωσή τους, που ζουν σε συνθήκες απαράδεκτες. Εάν δεν μπούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, λύση δεν μπορούμε να δώσουμε. Εμείς ως γυναίκες θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε τα πράγματα και να περιγράψουμε την κατάσταση που βλέπουμε στις χώρες μας. Και στην Αυστρία δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και στην Αυστρία έχουμε στους καταβλισμούς των προσφύγων το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε αξιοπρεπή κατάσταση στις γυναίκες πρόσφυγες αυτούς τους καταπλησμούς. Δεν υπάρχουν αρκετές ε, ε καμπίνες ε, ντους ή άλλα μέτρα και συνθήκες προσωπικής υγιεινής που να αισθάνονται αυτές οι γυναίκες άνετα και σε αξιοπρέπεια. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για την πραγματική κατάσταση της χώρας μου. Και θέλω κλείνοντας να πω ότι μόνο με μια αποτελεσματική πολιτική υπέρ της ειρήνης, στην οποία θα εμπλακούν και οι γυναίκες, μπορούμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτή την σοβαρότατη πολιτική κρίση που διέρχεται ο κόσμος. Χωρίς τις γυναίκες δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Χωρίς τις γυναίκες δεν μπορούν να υπάρξουν συνθήκες αξιοπρέπειας για τον άνθρωπο. Και δεν μπορούν να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτή είναι η έκκλησή μου προς τις γυναίκες πολιτικούς που είναι σήμερα εδώ σε αυτήν την αίθουσα, παρακαλώ δείξτε θάρρος, δείξτε παρησία, προσπαθήστε να μιλήσετε ξεκάθαρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζετε στις χώρα σας. Για να μην εγκαταλείψουμε τις γυναίκες στη μοίρα τους. Πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε, πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε ευκαιρία στις γυναίκες αυτές για μια, για ζωή αξιοπρεπή. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Μια ναι, και μας έχουν απομείνει μόνο λίγα λεπτά ίσα ίσα για να ακούσουμε τις δύο καλεσμένες μας. Θα ήθελα να δεχτώ το γάντι που μου πέταξε μία ομιλήτρια και που είπε ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να προβλέψουμε περισσότερο χρόνο. Θα το κάνουμε γιατί Όντω ένα τόσο σημαντικό σεμινάριο αξίζει μια ολόκληρη μέρα συζητήσεων για να έχουν το χρόνο πολύ περισσότεροι συνάδελφοι να μιλήσουν. Πάντως σας ευχαριστώ θερμά, θερμά που ήρθατε, που λάβατε μέρος, που μας μεταφέρατε τις θέσεις και τις ευαισθησίες των χωρών σας. Θα συνεχίσουμε το έργο, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία, γιατί όπως είπε και κάποια συνάδελφος, αυτό είναι το καθήκον μας, είναι η υποχρέωσή μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Ως πολιτικοί θύνοντες ε, ε, στα θεσμικά όργανα, αυτό το καθήκον και αυτή την υποχρέωση έχουμε. Δεν μπορούμε να γυρίζουμε την πλάτη και να διαφορούμε για αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία που θα προσπαθήσω να προφέρω σωστά το όνομά της, κυρία Ίγκυρτ Πόρτ, φαντάζομαι ότι το κατακρεούργησα δυστυχώς. Η κυρία Γκισλαντότυρ ε, εκπροσωπεί το Τμήμα Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών στην Τουρκία και είναι Γενική Διευθύντρια για την Κεντρική και Ανατολική Ασία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ και επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστώ την Επιτροπή Γυναικών και Ισών Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκδήλωση που οργανώσατε και βέβαια για την πρόσκληση που μου να συμμετάσχω εκ μέρους του οργανισμού που εκπροσωπού Είναι πολύτιμη η ευκαιρία που μου προσφέρατε να παρακολουθήσω τις εργασίες σας και βέβαια να επικυρώσω τα ευρήματα για την αξιολόγηση της προσφυγικής κρίσης ε, για τη Μακεδονία, για τη Σερβία και τα ευρήματα της έρευνας που κάναμε πέρυσι στις, ε, στα συνοριακά αυτά σημεία. Ο σχεδιασμός και η ενημέρωση από ό,τι βλέπουμε δεν μπόρεσαν να απαντήσουν στις ανάγκες των γυναικών ή να τις προστατεύσουν επαρκώς. Δυστυχώς αυτό από πέρσι μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει. Πρέπει επίσης να πω ότι με καταπλήσει το πόσοι βουλευτές ήρθαν ε, από ολόκληρη την Ευρώπη για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει μέχρι τώρα φωτιστεί επαρκώς. Ας είμαστε ειλικρινεί όταν μιλούμε για ισότητα ευκαιριών και χειρεφέτηση των γυναικών. Πολλά λόγια λέγονται, προγράμματα αναπτύσσονται, ομιλίες, γίνονται σχέδια και έργα ε, ανακοινώνονται, αλλά δυστυχώς όλα αυτά πάσχουν από υλοποίηση και βεβαίως αυτό ισχύει και για τις γυναίκες πρόσφυγες. Ελπίζω και βλέποντας σας εδώ μπορώ να πιστεύω νομίζω ε, ότι όντως θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία συζητήσατε. Οι γυναίκες λοιπόν αυτές είναι γυναίκες που έχουν διέλθει τέσσερα χρόνια πολέμου στη Συρία και περισσότερους ακόμα χρόνους πολέμου και συγκρούσεων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Πρώτη φορά ύστερα από την κίνηση της κρίσης τώρα, τον Ιανουάριο του 2016, οι γυναίκες και τα παιδιά ε, έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά προσφύγων που φτάνουν μέχρι τις ακτές της Ελλάδας. Γυναίκες και κορίτσια πέφτουν θύματα της βίας, ε, της σεξουαλικής, της βίας σχετικής με το φύλλο από τους άλλους ταξιδιώτες τους πρόσφυγες, από τους λαθροδιακινητές, από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, από τρομοκράτες. Αυξάνονται τα νούμερα των γυναικών προσφύγων, όμως δεν ενισχύεται περισσότερο η υπηρεσία που του προσφέρεται στον δρόμο για την προσφυγιά. Όπως είδαμε τη Δευτέρα, αντιθέτω, αντιμετωπίσουν μια όλο και πιο αρνητική, εχθρική, στρατιωτικοποιημένη αντιμετώπιση στον χώρο μεταξύ Ελλάδας και Μακεδονίας στα σύνορα, αλλά και στα στους αυτοσχέδιους καταβλισμούς όπως η παράδειγμα στο Καλέ. Γυναίκες και παιδιά που είναι τα πρώτα και κύρια θύματα των ένοπλων συγκρούσεων στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται. Γίνονται θύματα, πέφτουν θύματα βίαιων επιθέσεων ε, και ε, εμπλέκονται σε αντιπαραθέσεις βίες ακόμα και εκεί που θα πρέπει να τους προσφέρεται η προστασία στις 29 Μαρτίου. Λέει ο Μιλήτρια, είδαμε να πέφτουν θύματα και των δακρυγόνων. Προφανώς εννοείται Φεβρουάριο. 29 Φεβρουαρίου. Είναι αυτά λοιπόν τα πρώτα θύματα. Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των προσφύγων και των δυνάμεων ασφαλείας αποτελούν επίσης ένα λόγο ε, για ε, τροφοδότηση αρνητικής ορολογίας και λόγου από ξεφνοφοβικές ομάδες στην Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια πολύ έφλεκτη κατάσταση, μια κατάσταση η οποία δεν θα αργήσει να μετατραπεί σε πυρκαγιά. Το για τις γυναίκες και τα κορίτσια είναι μια όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. Στις χώρες ε, του δρόμου των Δυτικών Βαλκανίων βλέπουμε να αναλαμβάνονται μονομερώς μέτρα για έλεγχο συνόρων. Με βάση τη συνθήκη της, Γενέ, Γενέβης, το δικαίωμα στην προστασία σημαίνει δικαίωμα σε ατομική υποστήριξη και εξέταση του αιτήματο για άσυλο. Όπω ε, τόνισε στι 26 Φεβρουαρίου ο Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, οι νέοι περιορισμοί δεν είναι συμβατή με τη συνθήκη του 1951 της ε, Γενέβης και αντίστοιχα του πρωτοκόλλου του 1961 ε, για την προστασία των προσφύγων. Γιατί πρέπει να γίνεται ατομικά η αξιολόγηση των αραγκών κάθε ετούντος του ασύλου. Η κατάσταση στα ελληνικά σύνορα επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Εχθές επιβεβαιώθηκε πως η Ελλάδα επαναπατρίζει στην Τουρκία, ε, επιστρέφει στην Τουρκία, επαναπροωθεί στην Τουρκία 308 ε, πρόσφυγες, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με τη συνθήκη επαναπροώθησης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξαίρεση για την προστασία των ανθρώπων που έχουν θύματα ιδιαίτερος ε, παραβιάσεων των δικαιωμάτων, όπως πρόκειται για γυναίκες, όταν πρόκειται για γυναίκε οι οποίε έχουν υποστεί σεξουαλική βία ή ε, ΛΟΑΔΜ που κινδυνεύουν από διώξει όταν επιστρέφουν στι πατρίδε του. Εδώ βλέπουμε ότι θα πρέπει και η συμφωνία τη Κωνσταντινούπολη, σχετική συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, να γίνεται σεβαστή και από τη Σερβία για να προσφέρονται οι σχετικέ υπηρεσίε και το άσυλο στου πρόσφυγε, όπω ε, προτείνεται και από το σχέδιο εκθέσεω για την κατάσταση των γυναικείων προσφύγων και του ε, άσυλο. Ο κίνδυνος σεξουαλική βία, καταναγκαστικούς γάμους, ε, ε, γενετική λιτεροδεκτομή και άλλα τέτοια, άλλες τέτοιες ασκήσεις, ε, εκδηλώσεις βίας κατών γυναικών πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένη αναγνώριση του δικαιώματος σε άσυλο. Πρέπει να υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιολόγηση με βάση το κριτήριο και του φύλου του ασύλου Πρέπει να προσφέρεται νομική αρρωγή στις γυναίκες που αιτούνται άσυλο και πρόσφυγες, πρόσβαση σε γυναίκες διερμηνείς, υποστήριξη περιγενετική, υποστήριξη σχετική με τα παιδιά, δυνατότητα για ε, διατύπωση ε, αυτόνομου αιτήματο ασύλου χωρίς να δεσμεύεται από τον σύζυγο η αίτηση του δικαιώματος ε, σε άσυλο της γυναίκας, όπως πολύ σωστά λέει η έκθεσή σας. Γιατί πολλές φορές αυτό το δικαίωμα περιορίζεται από την επιλογή του συζύγου και γι' αυτό θα πρέπει το δικαίωμα αυτό να αναγνωρίζεται αυτόνομα στις γυναίκες. 2,5 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες είναι στην Τουρκία στην οποία εγώ εργάζομαι, μισές είναι γυναίκες της ε, Περισσότερε έχουν εγκαταλείψει άντρε του οι οποίοι έχουν ήδη πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρουν θέσει εργασία και τώρα είναι όλο και πιο δύσκολη δυνατότητα επανένωση των οικογενειών και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερε είναι οι χώρε οι οποίε ε, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιορίσουν το δικαίωμα στην επανένωση. Η Δανία, η Γερμανία και άλλε χώρε ίσω να ακολουθήσουν. Και κλείνοντα, δεν ήθελα να πω ότι στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είναι αδύρυτη πλέον η ανάγκη να εκφραστεί μια γενική πολιτική βούληση, να εκδηλωθεί πολιτικό θάρρο. Χρειαζόμαστε πολιτικού που θα έχουν τη βούληση να αναπτύξουν ένα φιλόδοξο και γενικό, ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματο, τη υποδοχή των προσφύγων, με τρόπο ανθρώπινο και αξιοπρεπή. Θέλουμε πολιτικού οι οποίοι θα μπορέσουν να αναλάβουν βήματα και να επιδείξουν αλληλεγγύη και να αντιμετωπίσουν και τις προκαταλήψει και το μίσος, να δώσουμε μια χείρα βοήθεια στις αδέλφια μας αυτά που κινδυνεύει η ζωή τους, που κινδυνεύει η αξιοπρέπειά τους και τα ανθρώπινα τους δικαιώματα πάνω στις αξίες τις οποίες εξτηρίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται πολιτική βούληση και η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του φύλου που σήμερα καταγράφηκαν στη σημερινή συνεδρίαση ώστε να ληφθεί και το επόμενο βήμα και στην προσεχή σύνοδο Ευρώπης-Τουρκίας εδώ τη Δευτέρα στις ε, Βρυξέλλες να επι... σημανθούν τα αισθήματα αυτά και όπως είπε και ο Μάρτιν Σούλτς πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εναρκτήρια παρέμβασή του και γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που με υποδεχθήκατε εδώ και εύχομαι Όπω είπα, να πραγματοποιηθεί το επόμενο βήμα και να περάσουν τα θέματα αυτά και στη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία Δευτέρα. Σα ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μέρι Χόνιμπολ, που είναι ευρωβουλευτή και η συγγήτρια, όπως ξέρετε, τη έκθεση που εγκρίναμε ήδη στην Επιτροπή Δικαιωμάτων τη γυναίκα και την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των γυναικών που ζητούν άσυλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την τεράστια προσπάθεια που έκανε επαφή με τι οργανώσει και την έρευνα που έκανε προκειμένου να εξοικειωθεί με την πραγματικότητα και προσπάθησε και να συμφιλειώσει και τις ε, διάφορες πολιτικές απόψει, ώστε να ακουστεί μια ενιαία και συμπληρωμένη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. Κυρία Χόνιμπολ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την παρουσία μου εδώ και για την ευκαιρία που έχω ως εισηγήτρια αυτής της πολύ σημαντικής ε, υπόθεσης, αυτού του πολύ σημαντικού θέματο να σα πω δύο λόγια και να μιλήσω για λίγα δυστυχώς ε, από τα πράγματα που ακούσαμε σήμερα, γιατί δεν έχουμε χρόνο για όλα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και σας ευχαριστώ γιατί μας τιμήσατε με την εμπειρία και τις γνώσεις σας. Και ε, έχω εντυπωσιαστεί που τόσο πολλοί συνάδελφοι και από τις εθνικές βουλές έκαναν, μπήκαν στον κόπο και ήρθαν σήμερα στις Βρυξέλλες και η συμβολή όλων ήταν πραγματικά ε, πολύτιμη. Θα ήθελα να απηχήσω αυτό που είπε η κυρία Γεσλαντότηρα, ότι χρειαζόμαστε πολιτικό θάρρος και πολιτική βούληση. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και φαίνεται και εξαιρετικά δυσεπίλητη. Αλλά αν ανασκομποθούμε και συνεργαστούμε, πιστεύω ότι θα βρούμε λύση. Αυτό που αναζητούμε σήμερα είναι μια λύση για να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών σε αυτή τη σύγκρουση ε, και να, κάνουμε, να βελτιώσουμε κάπως την κατάστασή τους. Και φυσικά από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ε, από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε στη συζήτηση. Και φυσικά όλοι, και οι γυναίκες και τα παιδιά, αξίζουν σωστής ε, ανθρώπινης μεταχείρισης με βάση τις αξίες και τις αρχές μας. Και φυσικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ειδικέ ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών και το πόσο περισσότερο ευάλωτες είναι. Ε, δυστυχώς ε, δεν έχουν ληφθεί υπόψη αυτές οι ειδικέ ανάγκες και η ευπάθεια τροτότητα των γυναικών και των κοριτσιών που πραγματοποιούν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη, αλλά όπως ακούσαμε, η προοπτική του φίλου, η σκοπιά του φίλου, η... τα δεινά που παίρνουν οι γυναίκες, οι οδύνες τους, αυτά που αντιμετώπισαν δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά στην κοινή γνώμη. Δεν φαίνονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Πιστεύω όμως ότι και με τη σημερινή εκδήλωση και με την έκθεση διορθώνουμε κάπως αυτή την κατάσταση ε, την ε, τρίτη ευκαιρία της Παγκόσμιας ε, ημέρας των γυναικών θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια. Καταφέραμε να μπει στην ημερήσια διάταξη τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα γιατί είναι συμβολική η συζήτηση αυτή ακριβώς τη μέρα και η ομάδα, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών Θέλουμε να αναδείξει τη σημασία που έχει σε αυτή την Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα το ζήτημα των γυναικών προσφύγων και του άσυλο. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διάσταση του φύλου σε όλο αυτό το ζήτημα. Και επίση να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση και τι κυβερνήσει των χωρών μελών και οι χώρε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τη υποδοχή των προσφύγων ή και τι χώρε προορισμού των προσφύγων ε, τι ενθαρρύνουμε και τι ευσυχώνουμε να αναλάβουν δράση. Έχουμε πολύ έργο μπροστά μας και εμείς ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να φροντίσουμε και οι δικές μας κυβερνήσει, να μην φυστούν προσπαθειών ώστε να αντιμετωπίσουν ε, συνολικά το πρόβλημα των γυναικών προσφύγων. Γιατί διανύουμε και πολιτική κρίση, όχι μόνο προσφυγική. Και πολλοί επισήμαναν την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες αυτής της κρίσης, τα αίτια αυτής της κρίσης. Γιατί ε, τόσο πολλοί πρόσφυγες ε, ξεριζώνονται από τις αιστείες τους και έρχονται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει η ανάλυση αυτών των ε, αιτίων να γίνει τμήμα της εξίσωσης για την αναζήτηση λύσης. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρούμε λύση, αλλά ακόμη συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές. Και φυσικά συμφωνώ με την έκκληση για την ειρήνη, γυναίκες και ειρήνη. Ε, οι, περισσότεροι, οι περισσότερες ακτιβίστριες για την ειρήνη είναι γυναίκες ε, και οι φεμινιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη δίνουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στο θέμα της ειρήνης. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και στην προσφυγική κρίση, να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη της ειρήνης. Όπως ακούσαμε, η κρίση η προσφυγική γίνεται κρίση για τις γυναίκες, γιατί αυξάνονται οι οι αριθμοί των γυναικών έχουν ξεπεράσει πια το 50% των προσφύγων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση πια τα, οι στατιστικές. Μας τα είπε και η UNICEF. Για πρώτη φορά το 60% των προσφύγων είναι πια γυναίκες, ενώ πέρυσι ήταν μόνο 20%. Ε, και έχει αυξηθεί εντυπωσιακά και ο ρυθμός των παιδιών Οπότε θα πρέπει να εγγύψουμε και σε αυτό το ζήτημα, γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι αυτή η τάση θα παραμείνει ανωδική. Επίσης, πολλοί ε, ζήτησαν να δώσουμε το λόγο στις ίδιες τις γυναίκες πρόσφυγες και χαίρομαι που είχαμε μία πρόσφυγα από το Ιράκ που μας μίλησε σε ένα από τα εργαστήρια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή των προσφύγων γυναικών γιατί ακούσαμε πολλά από τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τις ε, οργανώσεις που παρέχουν συνδρομή στους πρόσφυγες, αλλά καλό θα ήταν να ακούσουμε και τις μαρτυρίες και τα προσωπικά βιώματα αυτών των γυναικών. Των γυναικών που εγκατέλειψαν τις αιστείες τους, άφησαν το σπιτικό τους και ξεκίνησαν ιδιαίτερα επικίνδυνα ταξίδι, ε, μερικές φορές και με τα παιδιά τους, αντιμετωπίζοντας βία καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, βία από τους άλλους πρόσφυγες, βία και από τις ε, αρχές υποδοχής ή διέλευσης και αντιμετώπισαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και αντίξωες. Είναι σχεδόν ασύλληπτο πόσο, πόσα δεινά περνάνε αυτές οι γυναίκες. Και δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, αλλά αν έχετε παρακαλώ ε, επισκεφτείτε το Παρλαμεντάριου ε, και έχουμε μια έξεση φωτογραφίας ε, της φωτογράφου Μαρή Ντρινιέ έγινε αυτή η έκθεση με την οργάνωση της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σας δίνει μια εντύπωση της κατάστασης. Ε, γυναίκες που αφήνουν τα σπίτια τους αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Νομίζω ότι έχουμε καθήκον να τους δώσουμε μια ελπίδα για το μέλλον. Τέλος ήθελα να ευχαριστήσω του τους διοργανωτές, να ευχαριστήσω τα, όσους ε, έλαβαν μέρος τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Γραμματεία για την ε, ε, ανεκτήμητη συνδρομή και πιστεύω ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε την εκστρατεία ε, ζητώντας καλύτερη ζωή και δικαιώματα για τις γυναίκες πρόσφυγες και παιδιά πρόσφυγες. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάνιμπολ. Να ευχαριστήσω και τη διερμηνία που μας έδωσε πέντε λεπτά επιπλέον για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το σεμινάριό μας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συμμετοχή σας και να σας πω ότι ε, μετά το πέρας αυτής της εκδήλωσης, ε, αφού τελειώσαμε δηλαδή, ε, έχουμε μία μικρή δεξίωση στην, στην άλλη πλευρά του κτηρίου, στο Γενοντή Μενουχήμ και να σας ζητήσω να πάμε όλοι μαζί για να μην χαθούμε εδώ πέρα γιατί είναι μεγάλες αποστάσεις. Ευχαριστώ.